Σας καλώ, συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι βουλευτές, να ψηφίσουμε επί του ψηφίσματος που αναφέρεται στη σύναψη της συμφωνίας με την Γεωργία. Τροπολογία 1, Δυνατάσιος. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε. Ε, καταπίπτει η 5, παράγραφος 15. Εδώ έχουμε... Η, η 5 καταπίπτει, διότι ανακρύφει η 1. Παράγραφος 15, αντίστοιχες τροπολογίες. Ε, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να το ε, ε, ηλεκτρονικό έλεγχος ψηφίζουμε για την 26. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. Ο κ. Πρέντα, ε, περί προφορικής τροπολογίας. Κύριε Πρέντα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω αυτή την προφορική τροπολογία, αλλά πρώτα-πρώτα θέλω να χαιρετήσω τον Μιχαήλ Σακασβίλη, τον προηγούμενο τέος πρόεδρο της Γεωργίας, που και αυτός παρίσταται. Και θα ήθελα να καταθέσω μια προφορική τροπολογία, μια νέα παραγραφή υπαριθμών 10, 6. Θα έχει ως εξής. Χαιρετίζουμε τον ε, Σάζη με Επιτροπή Παρατήρησης του Δεκεμβρίου και επίσης απευθυνούμε έκκληση προς την κυβέρνηση της Γεωργίας να καταβάλει προσπάθειες ούτω ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρόεδρε, ε, υπάρχει ένσταση για αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφίζουν την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία. Τροπολογία υπαρθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρασε And it is adopted. Εγκρίνεται. The last vote is on the report τελευταία δηλαδή, ψηφοφορία είναι η, η έκθεση Μαμπίκιν όσον αφορά την Συμφωνία Σύνδεση ε, Ένωση και Γεωργία. Έχουμε ασκή ψηφοφορία, ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας. And it is adopted. Και εγκρίνεται. Thank you, colleagues. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι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 από τους πράσινους ένα αίτημα για το διορισμό του κυρίου Έρνεστ Μαραγκάλ σαν ε, μέλος της Επιτροπής